Okay, we we can start, yeah. Good morning, colleagues. Let's start our job. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε την ε, κοινή συνεδρίαση έκων και γυναικών. Καταρχάς, θα ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει την ημερήσια διάταξη. Όχι εγκρίνεται ένα μόνο σημείο. Πολιτικές ισότητας και φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέταση των τροπολογιών. Συζητούμε σήμερα τις 189 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για την κοινή έκθεση για την ισότητα των φύλων και τις πολιτικές, ε, τις φορολογικές. Μαρίσα Ματίας από την ΕΚΟΝ και Ερνέστο Ούρτασούν από την Επιτροπή των Γυναικών είναι οι συνεισηγητές μας και θα ακούσουμε τις ε, θέσεις τους στα κύρια σημεία της έκθεσης και των τροπολογιών και ε, τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Ματίας να λάβει το λόγο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσω με ευχαριστίες προς τους σκιώδεις συγητές και τον συνεισηγητή για τις τροπολογίες τους και να σας ενημερώσω ότι ήδη είχαμε μια πρώτη συζήτηση για τις 189 αυτές τροπολογίες και τη συζήτηση κάποιων συμβαστικών τροπολογιών που ήδη έχουμε εκπονήσει και καλύπτει μεγάλο τμήμα των, τροπολογιών. Πάντω ε, ήταν πολύ επικοδομητικό το πνεύμα όλων των συναδέλφων και του ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Και υπάρχει μια σχετική βούληση να καταλήξουμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Γιατί είναι Πραγματικά πολύ σημαντικό και συμφωνούμε με τον συνεισηγητή τον κύριο Ορτασούν ότι θα πρέπει το θέμα της ισότητας των φύλων να το φέρουμε στο επίκεντρο της χάραξης των φορολογικών πολιτικών. Γιατί είναι μείζον ζήτημα. Και μπορεί να φαίνομαι υπεραισιόδοξη, αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες που θα καλύπτουν τις ε, πολυάριθμες τροπολογίες. Ε, ένα θέμα που έμεινε κρεμές και θα πρέπει να το κανονίσουμε είναι το θέμα της φορολόγησης και κυρίως ε, της εξατομικευμένης φορολόγησης, της υποβολής δηλαδή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων στον οικοκύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα και καλό θα ήταν να το συζητήσουμε. Φαντάζομαι οι συνάδελφοι μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα θέματα της έκθεσης, ε, αν προτιμάν, αλλά νομίζω καλό θα ήταν, ε, ε, μια και έχουμε την ευκαιρία, να συζητήσουμε κυρίως αυτό το θέμα της ατομικής φορολόγησης και να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε συμβαστική λύση για αυτό το θέμα της ατομικής φορολόγησης, γιατί εξακολουθεί να είναι από τα κεντρικά σημεία της έκθεσης αυτό το ζήτημα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων για να δω αν μπορούμε να βρούμε κάποια λύση για ένα από τα κεντρικά ζητήματα της έκθεσης, το θέμα της ατομικής φορολόγησης. Σας ευχαριστώ κυρία Ματίας. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ουρτασούν. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Το ενδιαφέρον ε, για την έκθεσή μας ε, ήταν πολύ ζωηρό Εξού και η πληθώρα των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Πιστεύω ότι θα είναι καλό το κείμενο και ένα καλό βήμα προόδου για να καθοδηγήσει τις δημόσιες πολιτικές για την ισότητα φύλων και τη φορολογία. Και αν το εγκρίνουμε, πραγματικά θα έχουμε ένα πολύ καλό κείμενο για, για τα θέματα αυτά και μπορούμε να ε, επηρεάσουμε όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τις ειδικές συστάσεις χώρα, αλλά και τις πολιτικές των κρατών μελών. Ε, Γενικώ πάντως και παρά τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών, ήδη από την πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών διαπίστωσα μεγάλη επιθυμία για ανέβρεση συμβαστικών προτάσεων. Καταρχήν θα πρέπει να προσαρμόσουμε την άμεση και άμεση φορολογία στην ισότητα των φύλων, να εξορθολογήσουμε τις συστάσεις ε, ε, για τη φορολογική πολιτική συνεκτιμώντας τη διάσταση του φύλου και παρά κάποια συντακτικά σημεία που τα διορθώνουμε, διαπίστωσα στην πρώτη συνεδρία στο σχεδόν εισηγητών ότι η πλειοψηφία των ε, πολιτικών ομάδων ε, είναι υπέρ της ανέβρεσης συνένεσης. Μία εκκρεμότητα έχει μείνει το θέμα της εξατομίκευσης της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή της υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογικών. Ε, κατά τη γνώμη μου, το ελάχιστο που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση είναι ότι θα πρέπει να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να πατάξουν ε, οποιαδήποτε διάκριση προκύπτει ε, από την κοινή φορολόγηση, από την υποβολή δηλαδή ενιαίας φορολογικής δήλωσης. Γιατί μερικές φορές έχουμε διακρίσεις λόγω αυτής της κοινή φορολόγησης. Τώρα, αν θα πρέπει να απευθύνουμε σύσταση για ατομική φορολόγηση στα κράτη-μέλη, να βρούμε μια χρυσή τομή, αυτό θα το συζητήσουμε στην πορεία για να βρούμε μια συνενετική λύση. Πάντως θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα βρούμε μια λύση, προκειμένου να έχουμε μια έκθεση που θα τύχει θερμής υποστήριξη στην Επιτροπή. Αυτή είναι η δεδηλωμένη βούληση και των δύο συνεισηγητών της Μαρίας και εμού. Ευχαριστούμε κύριε Ορτασού. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ομίγυρη. Θα ξεκινήσω βέβαια από τους κοιόδης ηγητές και πρώτα απ' όλα από τον κύριο Γκέρχολτ που αντικαθιστά ένας άλλος κοιόδης ηγητή. Ε- Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έλαβα ορισμένε σημειώσει ε, χθε, είναι στα αγγλικά. Κυρία Χάιση και κύριο Σάβο, ε, ζητούν συγγνώμη που δεν είναι εδώ σήμερα το πρωί. Όμως ε, ήθελα να σας παρουσιάσω τις θέσεις ε, του ΕΛΚΑ για αυτή την έκθεση. Πάνω από 70 τροπολογίες ε, κατέθεσε το ΕΛΚ για αυτή την έκθεση. Γι' αυτό δείχνει ότι εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε επικοδομητικά σε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε μία ε, αρκετά παραγωγική συνεδρίαση των συντονιστών μέχρι τώρα και νομίζω ότι ε, μπορούμε έτσι εγκαίρως να ολοκληρωθεί το έργο για αυτή την έκθεση. Να επισημάνω ορισμένε βασικέ προτεραιότητε για αυτή την έκθεση, παρότι αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν ζητήματα έμεσων, έμεσων διακρίσεων μέσω φορολογικών πολιτικών, θεωρούμε ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να ε, εξετάσουμε ε, τα ζητήματα της αγοράς εργασίας. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και η σωστή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Η φορολογική πολιτική γενικά ε, έχει έναν χαρακτήρα ή πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα ουδέτερο ως προς το φύλλο. Ε, φυσικά οι πολιτικέ στην αγορά εργασία, οι εργατικέ πολιτικέ είναι αυτέ που μπορούν να δημιουργήσουν διακρίσει. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τονίζουμε επίση ότι τα φορολογικά συστήματα είναι ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μπορούμε να του ε, παροτρύνουμε να εξετάσουν και να λύσουν ή να πατάξουν τυχόν διακρίσει στα κοινά φορολογικά ζητήματα, όμως εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, μονομερή κριτική ενός συγκεκριμένου φορολογικού συστήματος έναντι άλλου. Δεν μπορούμε επίση να επιβάλλουμε συγκεκριμένε λύσεις ή να μην τηρήσουμε και την ε, ελεύθερη επιλογή που έχουν ε, οι οικογένειες στην Ευρώπη να επιλέξουν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ελεύθερη επιλογή, η ελεύθερη επιλογή για τους Ευρωπαίους πολίτες σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ και τον λεγόμενο ροζ φόρο, θεωρούμε ότι η διατύπωση είναι προβολική και θα πρέπει να ε, το κείμενο. Αυτά θα πρέπει να λυθούν ε, στην οδηγία για τον ΦΠΑ και η πρόσφατη ε, πρόταση για τους συντελεστές ΦΠΑ δίνουν περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη να θέσουν ακόμα και μηδενικό φόρο ε, για προϊόντα υγιεινής. Συνεχίζονται λοιπόν ε, οι διεργασίε. Ε, εκτιμούμε το ανοιχτό πνεύμα των εισηγητών, ε, φυσικά τελικά πρέπει να δούμε και ε, τους τελικούς συμβιβασμούς και κάποια ζητήματα που εκκρεμούν στην έκθεση. Το ΕΛΚ προσβλέπει στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπερές παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εισηγητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά όταν ε, βλέπει κανείς ε, τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν πολλές τροπολογίες και νομίζω ότι υπάρχει υλικό για να έχουμε μια πολύ καλή θέση των δύο επιτροπών σε έναν τομέα ε, που προσφάτως μόνο ανέλαβε να εξετάσει το Κοινοβούλιο. Ο τελικός στόχος είναι ε, να αναδείξουμε ε, τις έμεσες τρευλώσεις και διακρίσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στα κράτη-μέλη που ε, λειτουργούν τιμωρητικά προς τις γυναίκες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας, που είναι κέριο ζήτημα, προκειμένου εκείνες να μπορούν να διάγουν έναν ανεξάρτητο βίο από πλευράς πόρων η δίκαιη φορολόγηση ανδρών και γυναικών, ε, ιδίω ό,τι έχουν να κάνουν με τα νοικοκυριά, ε, όπου βλέπουμε ότι πλέον η επιστροφή της γυναίκας στην αγορά εργασίας ε, δεν συμφέρει οικονομικά το ζευγάρι. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Δεν πρέπει όμως αυτό να αποβεί σε βάρος των πλεονεκτημάτων που δίνουμε στα ζευγάρια για λόγους δημογραφικούς περισσότερο σε ορισμένα Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τη φορολογία για να βελτιώσουμε τις ε, υποδομές υποδοχή παιδιών, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί είναι ένας ε, τρόπος αντιστάθμισης αυτής της εξατομίκευσης ε, των φόρων και να επιτρέψουμε στις γυναίκες πιο εύκολα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, σε ε, μια πρόταση που θα διαβάσω στα αγγλικά, όμως ε, προσπαθεί να επιλύσει ένα από τα βασικά εκρεμή ζητήματα. Σε ό,τι αφορά ακριβώς ε, την προσωποποίηση της φορολόγησης. Παροτρύνουμε λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην εξοδικευμένη φορολόγηση, ενώ θα διασφαλίζουν την το πλήρη σεβασμό όλων των άλλων πλεονεκτημάτων που συνδέονται με την γονεϊκότητα στα σημερινά φορολογικά συστήματα. Αυτή είναι μια προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Νομίζω ότι η έκθεση μέσω των συμβαστικών λύσεων θα υποστηρίξουν όλα τα κρατημέλη που υπό το καθεστώς της αναθεώρησης ε, της οδηγίας για το ΦΠΑ ε, θα εξετάσουν εκ νέου τον, ε, το pink tax, τον ροζ φόρο και είναι θεμελιώδες ζήτημα η τροφοδότηση ε, αυτού του ζητήματος ότι φορά την συλλογή πληροφοριών και να μελετήσουμε τον αντίκτυπο των δημοσιονομικών και φορολογικών πολιτικών ε, που διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, για να στοχεύσουμε καλύτερα ε, την ε, προλική μας πολιτική. Καλή δύναμη. Εύχομαι στους δύο συνεισηγητές. Ευχαριστούμε κυρία Μπέρες. Και τώρα λόγω στον κύριο Τρεμόσα από τους Φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές για το έργο τους. Εμείς οι φιλελεύθεροι αντιμετωπίζουμε πια μια νέα πραγματικότητα. Έχουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις ανισότητας στα κράτη-μέλη και στους διάφορους τομείς και μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Θα πρέπει όμως να δούμε ποια είναι και τα καταναλωτικές ε, συμπεριφορές ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που αγοράζουν, γιατί δεν αγοράζουν τα ίδια προϊόντα άνδρες και γυναίκες στις αγορές, είτε για ζητήματα υγείας ή υγιεινής, αλλά και άλλα. Και αν υπάρχει ε, απόδειξη ότι υπάρχει προκατάληψη στη φορολογία και μεροληψία εις βάρος των γυναικών σε ό,τι αφορά αυτό το καλάθι των προϊόντων, των αγαθών που αγοράζουν άνδρες και γυναίκες, θα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι προς τη νέα πραγματικότητα και αν αποδειχθεί αυτό να γίνει μια προσαρμογή των δημόσιων πολιτικών προκειμένου να ασπαστούν τη νέα πραγματικότητα. Δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση μεταφορών κονδυλίων, αλλά μια ένωση βέλτιστων πρακτικών. Και με την άποψη του ΕΛΚΟ ότι σίγουρα η φορολογία εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα αρμοδιότητα εθνική. Βέβαια, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλουμε τις βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθούν τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τους στόχους τους για περισσότερη ισότητα και πιο ισορροπημένο αντίκτυπο της φορολογίας ε, με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου. Γι' αυτό και οι φιλελεύθεροι θα φροντίσουν να διευκολύνουν τη συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να δώσουμε συστάσεις στα κρατημέλη για να βελτιώσουν τις φορολογικές τους πολιτικές. Ευχαριστούμε κύριε Τρεμόσα. Άλλος κανείς παρακαλώ. Η κυρία Τζούλι Βόρτ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι ιδιαίτερα αρμόδια για το θέμα αυτό, αλλά επειδή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της ισότητας για τις γυναίκες, η ισότητα μεταξύ των φυλών έχει πολύ μεγάλη σημασία και οτιδήποτε κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατρέχεται από τα θέματα της ισότητας των φύλων. Οπωσδήποτε και η φορολογία έχει τη σημασία της, έχει ψηλή σημασία σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι όταν δεν αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο οι γυναίκες, το τίμημα το πληρώνει η ολόκληρη κοινωνία συνέπειες υπάρχουν από την έλλειψη ισότητας, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένουμε. Και σε αυτό μπορώ να καταλογίσω και την βία. Μια κοινωνία η οποία δείχνει γνήσιο σεβασμό στις γυναίκες, προσφέρει ισότιμες ευκαιρίες σε κάθε τρόπο, σε κάθε μορφή ε, και τομέα της ζωής. Νομίζω ότι έχει διαφορετική εικόνα γιατί υπάρχει πάντα ένας σχετισμός και συνάφεια ε, ως προς τη βία που υφίστανται οι γυναίκες και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζει η κοινωνία. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να ε, μεριμνήσουμε ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Είχα σε ένα κομμάτι αρμοδιότητα για την έκθεση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης και κοιτώντας το θέμα της οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτονομίας των γυναικών διαπιστώσαμε ότι και ειδικά για τις γυναίκες με ε, δυσκολίες ή με αναπηρία η λιτότητα είχε καταστήσει τόσο δύσκολη την καθημερινή ζωή, το να ανάψουν το καλοριφέρι, να βάλουν ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι για τα παιδιά τους. Όλα αυτά νομίζω πρέπει να τα λύσουμε και μέσω των φορολογικών πολιτικών, γιατί πολλές είναι γυναίκες που πλήττονται από μέτρα ε, εφόσον δεν υπάρχει η μέρημνα για την ισότητα. Με τους συναδέλφους λοιπόν θα κοιτάξω να έχουμε μια καλύτερη και πιο ισότιμη μεταχείριση, πιο δίκαιο κόσμο και για τις γυναίκες και τις οικογένειές τους ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ τους συνεισηγητές να λάβουν το λόγο. Τώρα κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ και πολύ σύντομα γιατί θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Αναφέρθησαν όλοι σε κέρια ζητήματα, σε σοβαρά και σημαντικά ζητήματα. Οπωσδήποτε δεν έχουμε στόχο να παρισφρήσουμε στις ε, δικαιοδοσίες, στις φορολογικές των κρατών μελών. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση, ούτε και πρόκειται να υπάρξει. Αλλά κοινέ πολιτικές με έμεση, έμεσο αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων, μπορούν να άπτονται και τη φορολογική πολιτική. Εάν υπάρχει ένα κοινό σύστημα ΦΠΑ, παραδείγματι, και αν δούμε ότι υπάρχουν κάποια μοντέλα κατανάλωσης που σχετίζονται με το φύλλο, οπωσδήποτε έχουμε δικαίωμα να το εξετάσουμε πώ αντιμετωπίζουν την ισότητα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Δηλαδή, εκεί όπου υπάρχουν κοινέ διαστάσεις, εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη ε, ανισότητα στην αντιμετώπιση των γυναικών, πρέπει εμείς να φροντίσουμε αυτό το χάσμα, αυτό το, αυτή η ανισορροπία να μην ενισχυθεί. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και ιδιαίτερα την Περβόνς για την ε, διατύπωση που προτείνει προκειμένου να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από το κύριο πρόβλημα που έχουμε κατά τη συζήτηση της έκθεσης. Συμβαστικά νομίζω είναι μια πολύ καλή πρόταση και βεβαίως μπορούμε να τη συζητήσουμε με όλους τους κοιόδης όταν έρθει η ώρα, αλλά είναι πολύ χρήσιμη και μπορώ να το πω από τώρα η συμβολή σου, Επίσης προς τον συνάδελφο για το ΕΛΚ που εκπροσωπεί δύο σκιώδεις, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις και τις, ε, τα μελήματα που εκφράζονται και βεβαίως διατυπώνουμε μια κοινή συμβιβαστική λύση στο τέλος με μέρημνα να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο προβλέπει η, η, νομική βάση μεν, αλλά εάν δούμε ότι δεν είναι η κατάλληλη νομική βάση, θα την αλλάξουμε. Γιατί εάν δεν φέρνει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, δεν κάνουμε τίποτα. Επομένως, θα καταθέσουμε τις προτάσεις και τις εναλλακτικέ λύσεις που θα εξασφαλίζουν με βάση την νόμιμη βάση που έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αν δεν προσφέρεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, θα κοιτάξουμε και να ζητήσουμε αλλαγή της νομικής βάσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ορτασούν εσείς. Όχι πρόεδρε τίποτε ιδιαίτερο, η Μαρίσα τα είπε όλα νομίζω. Απλώς θα σημειώσω ότι έχουμε κάθε βούληση για εξέβρεση μιας όσο το δυνατόν ευρείας συνένεσης. Ελπίζω πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα με όσο το δυνατόν λιγότερες ανατροπές. Ε, στο ζήτημα που έθιξε ο συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον φόρο στα ταμπών, όπως τον λένε, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Έχουμε όμως οπωσδήποτε ένα γνήσιο φαινόμενο άμεσης διάκρισης και, δια, και διακριτικής φορολόγησης σε πολλά κράτη-μέλη. Πολλοί έχουν ξεσηκωθεί στην Ευρώπη σε πολλές χώρες και ζητούν να ανατραπεί αυτό. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που εμένα με κινεί. Εδώ λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα διατυπώσουμε το κείμενο, πώς θα το ζητήσουμε, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να μπει στην έκθεση. Για την εξατομίκευση, η πρόταση της Πεγμός μου φαίνεται πολύ καλή. Ας ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν. Και ας δούμε αν το δέχονται και οι λοιπές ομάδες. Πάντως, καταρχήν, ε, η επιδίωξή μας θα είναι συνενετική λύση γύρω από την πρόταση της Περβάνς. Θα επιδιώξουμε, όπως έλεγα, στην προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών, των σκιωδών, να κλείσουμε το θέμα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κοινή συνεδρίαση 21 Νοεμβρίου για να ψηφίσουμε. Κοινή συνεδρίαση ΦΑΜ και ΕΚΟΝ τώρα έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις 9 ξεκινάει η ΕΚΟΝ.